Γιώργη Βοτολίπε, Τζάνταν Γεώργη Βοτολίπε, Γεώργη Βοτολίπε, έτρισε ο Ζηρώνη, Γιώργη Βοτολίπε, έτρισε ο Ζηρώνη. Έτρισε ο Ζηρώνη, Τζάνα μέτρισε ο Ζηρώνη, έτρισε ο Ζηρώνη, να Γιώργη Τούμα, έτρισε ο Ζηρώνη, να Γιώργη Τούμα μη βαρβίς Γιώργη, κατούσαμε κάτουσα μη βαρβίς να βοηνώ το πόλε, μη βαρβίς να βοηνώ το πόλε. Bravo, merci. Et notre voyage nous mène à présent en République tchèque avec Christian et Wojciech.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 This, bring, this brings a great culture, cultural diversity to our, our school and our city by the channel, one of the, one of the five most important harbour in Europe. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons découvrir la Croatie avec Magda et Franjo.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 in the international open mind for the Union in a global Europe. Alone we go faster, but together we go farther. Thank you. Merci. Et maintenant, Dragos nous emmène en Roumanie. Bonjour, ça va